Τελείωσαν εδώ οι αγορεύσεις του ενός λεπτού. Έχω δύο ανακοινώσεις από την ομάδα των συντηρητικών. Έλαβα την ειδοποίηση ότι αντικαθιστά ο κύριος Μπασίρ, τον κύριο Καμάλ, ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών. Δεύτερη ανακοίνωση που έχω είναι ότι ο κύριος Γιώργος Κατρούγαλος ανέλαβε θέση στην